Präsident. La seduta è ripresa. Il processo... Συνεχίζουμε. Τα χθεσινά πρακτικά έχουν διανεμηθεί. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις θεωρούνται δεκτά. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής